αυτοί οι διορισμοί θα θεωρούν ε, εγκεκριμένοι. Έχετε λοιπόν ε, τα ονόματα στον φάκελό σας ε, τώρα. Η υπογραφή των νομοθετικών κειμένων που ενεκρίθηκαν σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία το... την Τετάρτη εγώ και το Συμβούλιο θα υπογράψουμε εννέα ε, πράξεις ε, σύμφωνα με τον οργανισμό 74. Ε, οι τίτλοι αυτών των πράξεων έχουν δημοσιευθεί και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά μας. Αυτά σε ό,τι φορά τις ανακοινώσεις. Περνάμε τώρα στο θέμα της τροποποίησης της μεστής διατάξεως για τη Δευτέρα.